Oh, good morning everybody. I'd like to start the meeting, but I have... Θέλαμε να αρχίσουμε τη συνεδρίαση, αλλά είναι παρούσες μόνο δύο από τις επτά πολιτικές ομάδες. Το λέω για τα πρακτικά. Now, this 20 minutes <clears throat> Πέρασε και οι 20 ξεκινάμε. Πρώτο θέμα. Ενημέρωση. Θα την κάνω εγώ. Κανείς δεν είναι από τους τέσσερις εισηγητές, οπότε θα την κάνω εγώ. Πώς προχωρούν οι τριμερείς διάλογοι. Πρώτον, ο κανονισμός για το ISDS κανονισμό χρηματοοικονομικής ευθύνης. Όπως ξέρετε, με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας, η Ένωση ανέλαβε την ευθύνη για την πολιτική επενδύσεων. Χρειάζεται λοιπόν να κατανείμουμε την, ε, τις ευθύνες μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών σε περίπτωση ε, διαφορών σε, ε, σε θέματα επενδύσεων ποιος θα πληρώσει τυχόν αποζημιώσει. Ήταν εξαιρετικά αμφιλεγόμενο θέμα, όπως αποδείχθηκε το ζήτημα αυτό. Υπήρξε κάποια πρόοδος επί Λιθουανικής Προεδρίας, όχι μεγάλη. Τώρα προσπαθούμε να συνεργαστούμε με την ελληνική Προεδρία στο θέμα αυτό. Οι συνομοθέτε ε, συμφώνησαν να ζητήσουν από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια πιθανή συμβαστική λύση. Χτες, από λάθο σας ενημέρωσα ότι το Κοινοβούλιο αποφάσισε ήδη να δεχθεί το πακέτο που πρότεινε η Επιτροπή. Δεν είναι σωστό αυτό, δεν το έχουμε συμφωνήσει το Κοινοβούλιο μελετά ακόμα η, η αντιπροσωπεία μας ε, μελετά ακόμα τη συμβαστική πρόταση που έχει υποβάλει η Επιτροπή. Ο κ. Ζαλεύσκη είναι ο εκπρόσωπός μας στην ομάδα αυτή και θα συνημερώσει για πιθανές εξελίξεις. Πρόκειται για ένα από τα θέματα που θα έπρεπε νομίζω να, να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος της θητείας μα γιατί αποτελεί ένα βασικό κομμάτι της νέας επενδυτικής πολιτικής της Ένωσης. Και είναι προβληματικό το ότι έχουμε ήδη διαπραγματευτεί και συνάψει επενδυτικές ε, συμφωνίες ή κεφάλαια επενδυτικά σε άλλες συμφωνίες, αλλά δεν είμαστε σε θέση να πούμε στους εταίρους μας ακόμα ποιος θα είναι υπεύθυνο στο μέλλον, αν υπάρχουν διαφορές σε θέματα επενδύσεων. Οι εταίροι μας έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι θα συμβεί στο μέλλον. Κατόπιν, δύο κανονισμοί υπάρχουν που έχουν ήδη έχουν συμφωνηθεί. Ο ένας αφορά για την Συμφωνία Ένωση Σερβία, Συμφωνία Σταθεροποίηση και Συνεργασία. Υπάρχει συμφωνία σε επίπεδο τριμερών διαλόγων ήδη από το Δεκέμβριο. Το ίδιο συνέβη και με τον κανονισμό παροχή ε, εμπορικών προτιμήσεων στην Μολδαβία στα θέματα ε, εισαγωγών κρασιού. Το κείμενο είχε ήδη υιοθετηθεί στην Ολομέλεια Κάτι άλλο σημαντικό που έχουμε πρόοδο στις ε, διαπραγματεύσεις είναι ο εφαρμοστικός κανονισμός. Σημαντικό νομοθετικό κείμενο για να επιτρέψουμε στην Επιτροπή να λάβει μέτρα εξ ονόματος της Ένωσης εναντί τρίτων χωρών. Συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο να ζητήσουμε από την Επιτροπή να υποβάλει συμβιβαστικές προτάσεις. Η Επιτροπή το έπραξε. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την συμβιβαστική πρόταση της Επιτροπής υπό μορφή πακέτου υπό τον όρο ότι θα, κάνει, θα πράξει το ίδιο και το Συμβούλιο. Από ό,τι φαίνεται το Συμβούλιο δεν είναι ακόμα έτοιμο γι' αυτό το μέλλον του κανονισμού αυτού έχει ακόμα ένα μεγάλο ερωτηματικό. Κανονισμός για τα θέματα διπλών χρήσεων. Συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση με τον κύριο Φιάλ υπεύθυνο από πλευράς μας. Από ό,τι βλέπω, δύο ντοσχέ είναι σημαντικά με αβέβαιη ακόμα έκβαση συνολικά. Σχόλια? Όχι. Αλλά λείπουν και οι συγκητές. Δεν υπάρχουν σχόλια. Σημείο 10. Πως η κατάσταση για την Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών Ένωσης Βιετνάμ. Ψήφισμα, πρώτος ψηφίσματος. Ο Τσιοζάχραντιλ είναι ο εισηγητής, λείπει. Έρχεται, μου, είπε στο κοινο... μου είπαν στο κοινοβούλιο. Να, να διακόψουμε ή να ακούσουμε την επιτροπή. but Joanna is not terrorist. Well, I'll make a pause for 15 minutes. Διάλειμμα ενός τετάρτου. Look, this is a committee made of parliamentarians. If parliamentarians are, are not... Κοιτάξτε, πρόκειται για κοινοβουλευτική επιτροπή, απουσία κοινοβουλευτικών μελών. Τι να κάνω, πρόεδρος είμαι, επέμεινα προς τις, προς τις ομάδες να ορίζουν ένα κοινοβουλευτικό υπεύθυνο ζητώντας ένα μήνυμο αριθμού βουλευτών παρόντων σε κάθε συνάντηση. Τι άλλο να κάνω. Ξέρετε, όταν κανείς δεν είναι στην ώρα του, για να φτάσει να είναι στην ώρα του θέλει πολύ προσπάθεια. Διάλειμμα λοιπόν. 15 λεπτών. Υπότιτλοι Okay. Να επαναλάβουμε τις εργασίες μας. Ο εισηγητής μας, κύριος ε, Ζαχράτηλ, έφτασε. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στην ε, εξέταση του σημείου 10 σχετικά με τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών Ευρωπαϊκή Ένωση Βιετνάμ. Αποφασίσαμε να συντάξουμε ένα σχέδιο ψηφίσματο. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή μα, τον κύριο Γιάνν Ζαχράντιλ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, ζητώ συγγνώμη από όλους ε, τους συναδέλφους που τους ε, ανάγκασαν να με περιμένουν. Δυστυχώς ε, πήρα μια πρωινή πτήση από την Πράγα στις Βρυξέλλες χωρίς να σκεφτώ ότι θα έπεφτα σε μποτιλιάρισμα. Τέλος πάντων, ανόητη σκέψη, με συγχωρείτε που άργησα παρόλα αυτά. Τώρα, το θέμα μας. Ως ε, μόνιμος για τις ε, διαπραγματεύσεις ε, με το Βιετνάμ για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών, θέλω να σας παρουσιάσω αυτό το σχέδιο ψηφίσματος που έχει ως στόχο να αναφέρει τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τις εν λόγω συνομιλίες οι συνομιλίες αυτές προχωρούν σε καλό ρυθμό μέχρι τώρα και ενδέχεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του τρέχοντος. Χαιρετίζω λοιπόν την πρόοδο των συνομιλιών μετά τους πρώτους πέντε γύρους και θέλω να συγχαρώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ενημερώνει σε τακτά διαστήματα την ομάδα μας από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Ελπίζω να συνεχίσει να μας ενημερώνει διότι αυτή η πρακτική είναι πολύ καλή και με τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων και με τους κοιόδης θα έχω συνεχείς επαφές και με τους άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία. Χαίρομαι επίσης που η Επιτροπή το Μάρτιο στην Ολομέλεια ε, θα προβεί σε δήλωση σχετικά με τις ε, συνομιλίες, με τις διαπραγματεύσεις αυτές. Θα μας παρουσιάσει δηλαδή την κατάσταση ε, που βρισκόμαστε πριν λήξει αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος. Για να συνοψίσω, αφού σας πω ότι είναι υποχρεωτική η γνωμοδότηση του κοινοβουλίου αυτό το θέμα, ποια είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, η ανάγκη, η έκφραση των συνομιλίων να είναι συμβατή με τους κανόνες και υποχρεώσεις του ΠΟΕ και θέλουμε επίσης να υπάρχουν πραγματικά ωφέλη για τις, ε, για τις αμβαλόμενα μέρη, βελτιωμένες εμπορικές ροές, δημιουργία θέσεων απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, θα πρέπει να καταργηθούν και τα δοσμολογικά και τα μετασμολογικά εμπόδια, mm. βέβαια επιτρέποντας ε, μια σχετική ασυμμετρία στον των αγορών σε ευαίσθητους τομείς ε, ή ήδη και από τις δύο πλευρές τρίτων και τα δύο συμβαλόμενα μέρη θα πρέπει να σέβονται το δικαίωμα ε, του άλλου μέρους να ρυθμίζει ε, τα περί παροχής υπηρεσιών. Και οι ρυθμίσεις βέβαια δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν ε, το διμερές εμπόριο με μη δικαιολογημένα μέτρα. Τέταρτον, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να έχουν κάποια μέτρα επίλυσης διαφορών, διαμεσολάβησης για να καταργούνται ρυθμιστικά εμπόδια εναρμόνιση της συμμόρφωσης προς τα διεθνή πρότυπα, είναι κάτι που πρέπει να προωθηθεί. Πέμπτον, ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει τα συμφέροντά της, αλλά όχι μόνο με στόχο την απελευθέρωση της εθνικής ε, μεταχείριση, αλλά θέλουμε να έχουμε ισότιμη μεταχείριση όλων των παρόχων υπηρεσιών και προϊόντων σε τομείς όπως τραπεζικός τομέας, ασφαλιστικός τομέας, λογιστική, νομικά θέματα, μεταφορές και άλλα. Και θέλουμε να υπάρχει επίσης υψηλή, υψηλή επίπεδο προστασίας καταναλωτών. Να είναι εναρμοσμένες οι πρακτικές μεταξύ των επενδυτών. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ένα δίκαιο ε, διαφανές επιχειρηματικό περιβάλλον και για τις ιδιωτικές και τις δημόσιες επιχειρήσεις και να υπάρχει όσο δεύτερο μεγαλύτερη κάλυψη στον τομέα των διαγωνισμών, των δημοσίων προμηθειών. Επίσης, πρόσβαση στις αγορές να σχετίζεται και με την εφαρμογή και επιβολή των ε, διανοητικών ή πνευματικών δικαιωμάτων και των υγειονομικών και φυτοϊγειονομικών μέτρων για την ποιότητα και 8 και τελευταίο για αυτή τη Συμφωνία Ελευθέρω Εμπορίου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένα δεσμευτικό κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο να αντικατοπτρίσει την δέσμευση ΕΕ και Βιετνάμ να προωθήσουν το σεβασμό, την τήρηση και επιβολή των εθνών ανθρωπιστικών δικαιωμάτων και βασικών πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών. Και αν υπάρχει καταστρατήγηση, να επιβάλλονται μέτρα. Αυτά είχα να πω. Βέβαια, μπορούμε να επεξεργαστούμε ακόμη περισσότερο το κείμενο αυτό σε συνεργασία με του κοιόδη εισηγητέ, με στόχο το τελικό κείμενο, ελπίζω τουλάχιστον να εγκριθεί στην Ολομέλεια του Μαρτίου του 2014. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά και συγχωρήστε με που άργησα. Let's listen τώρα. Από το ΕΛΚ. Ο κύριος Γκλάτφεντερ. Με ευχαριστώ. Η εικόνα που έχω είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό κείμενο και πολύ καλό σχέδιο. Συγχαρητήρια λοιπόν στον συνάδελφο συντάκτη. Τα σημαντικότερα θέματα καλύπτονται όλα στο κείμενο, ένα προς ένα. Περιλαμβάνουν σωστές προτάσεις και μία όθη προσέγγιση. Δεν πέφτει δε το κείμενο στην παγίδα να αναμένουμε μια συμφωνία ελεύθερης συναλλαγών γενική που σχετίζεται με άλλες συμφωνίες. Καλωσορίζω την έκθεση και την υποστηρίζω. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες ε, που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ε, και που θα αντιμετωπίσουμε αλλά και πάλι συγχαρητήρια στον συντάκτη. Μπέντ Λάγκη για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή πολλά βασικά σημεία έχουν ε, σωστά περιγραφή. Ε, με δύο θα ασχοληθώ πιο συγκεκριμένα και ίσως ε, να κάνω και μια κάποια προσπάθεια να τα αναδείξω περισσότερο. Το πρώτο είναι η προστασία των ζώων. Ξέρουμε ότι το Βιετνάμ είναι μία από τις χώρες όπου το παράνομο εμπόριο ζώων είναι πολύ ανεπτυγμένο. Είναι ιδιαίτερα ε, επίσης και σημείο όπου γίνονται διεθνείς τέτοιες πράξεις, όχι μόνο δηλαδή παράνομο εμπόριο ε, στην εσωτερική αγορά. Πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη και να υπάρξουν ε, συμφωνίες ε, για το θέμα αυτό. Από ό,τι φαίνεται το Βιετνάμ είναι διατεθειμένο να αποδεχθεί να είναι μόνιμο ε, θέμα στη συζητήση μας ε, η ευημερία των ζώων, αλλά προσπαθεί ε, να το εντάξει όλος ιδιαίτερος στο κεφάλαιο της βιωσιμότητας. Αλλά επειδή είναι πολύ σημαντική αυτή η οικονομική δραστηριότητα, θα πρέπει να μπει στον τομέα SPS, Εκεί να βάλουμε λοιπόν την ε, προστασία των ζώων. Αυτό δεν είναι και τόσο επαναστατικό. Στην συμφωνία με τη Χιλή και με την Κορέα εκεί το έχουμε βάλει. Θα ήθελα λοιπόν να το βάλουμε και ε, στη συμφωνία με το Βιετνάμ σε αυτό το τομέα. Το άλλο είναι ε, το κεφάλαιο 13, δηλαδή πώς θα διαμορφωθεί το κεφάλαιο για την βιωσιμότητα. Θεωρώ ότι οι διαπραγματεύσεις μέχρι στιγμής σε μεγάλο βαθμό περιορίζονται σε συζητήσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της Κομισιόν. Δεν υπάρχει κανένα διάλογος με την κοινωνία των πολιτών, τα συνδικάτα για παράδειγμα. Δεν έχουν καμία δυνατότητα συμμετοχής. Πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν και η φάση ε, εκπόνησης αλλά και εφαρμογής μετά τη συμφωνίας να συμπεριλάβει σε μεγάλο βαθμό τον κοινωνικό διάλογο, τα συνδικάτα, άλλες οργανώσεις ούτως ώστε η συμφωνία αυτή να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του πληθυσμού. Θα ήθελα να ενισχυθεί αυτό το σημείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Για τους πράσινους. Για Σκακέλε. Ακριβώς. Για μένα προς το συμφέρον του πληθυσμού πρέπει να γίνεται το εμπόριο. Αυτό είναι το θέμα κλειδί. Για μας τους πράσινους πρέπει να παίξουν ρόλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να είναι συστατικό στοιχείο. Δεν ε, αρκεί να το αναφέρουμε στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Πρέπει να είναι ε, σημαντικό στοιχείο ε, της όλης συμφωνίας, οποιαδήποτε συμφωνία δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό χρειάζεται ε, μελέτη επιπτώσεων που πρέπει να κάνει η Κομισιόν στα πλαίσια του σχεδίου δράσης για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι ιδιαίτερο αναγκαίο σε αυτή την περίπτωση του Βιετνάμ, γιατί έχουμε διαπιστώσει επιδείνωση της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων τον περασμένο χρόνο φυλακίζονται άτομα μόνο και μόνο γιατί ασκούν ε, το δικαίωμα λόγου που έχουν, την ελευθερία έκφρασης. Θα πρέπει λοιπόν ε, να εφαρμόζονται οι διατάξεις των ανθρώπινα δικαιώματα. Επειδή λοιπόν είναι τόσο σημαντικό στοιχείο οποιασδήποτε συμφωνίας, αυτό πρέπει να προωθήσει η Ένωση. Για μας είναι λοιπόν πολύ ουσιώδες να προωθήσουμε, να επιβάλλουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεύτερον, ως πράσινη. δεν θέλουμε να συμπεριληφθεί το ISTS αυτή τη συμφωνία. Υπάρχουν πάρα πολλές επενδύσεις στο Βιετνάμ και αυτή τη στιγμή ε, γίνονται αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών νομίμως. Θα πρέπει οπωσδήποτε οι δυτικές εταιρείε να ε, δεσμεύονται να εφαρμόζουν τις διατάξεις κατά τέτοιων πρακτικών. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει περιθώριο ε, να δράσει το Βιετνάμ. Δεν μπορούμε να του ζητήσουμε να τα φιλελευθερωποιήσουν όλα, να τα απελευθερώσουν όλα αμέσως. Είναι αναπτυσσόμενη χώρα, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις δικές τους ευαισθησίες. Θέλουμε να γίνουν ε, να υπάρξει περισσότερη ευημερία. Η απελευθέρωση λοιπόν δεν είναι το καλύτερο σε όλους τους τομείς. Πρέπει να τους δώσουμε γενναιόδορες μεταβατικές περιόδους. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, είναι δεσμευτική η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πρόβλημα είναι εάν στην πράξη εφαρμόζεται. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Επόμενος, Πολ Μέρφυ για, ε, για την ε, νοτική αριστερά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Δεν συμφωνώ με την κατεύθυνση της έκθεσης. Έχω την εντύπωση ότι αντιμετωπίζει το Βιετνάμ ως ανεπτυγμένη χώρα, ζητάει αμοιβέ δεσμεύσεις κτλ. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει πολύ πιο εκπεφρασμένη αναφορά στο θέμα των ε, δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αναφερόμαστε στι βασικέ συμφωνίε του ILO, του Διεθνού Οργανισμού Εργασία και λέμε ότι πρέπει να γίνονται σεβαστέ, αλλά στην πραγματικότητα οι συμβάσει αυτέ παραβιάζονται συστηματικά στο Βιετνάμ. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι υπάρχει δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων, ελευθέρων συνδικάτων, πραγματικών ανεξαρτήτων συνδικάτων. Υπάρχουν θέματα καταναγκαστική εργασία και πρέπει ακόμη να πούμε ότι οι πολυεθνικές από τις χώρες μας δεν είναι αθώες είτε από πλευράς ε, εξαγωγών είτε από πλευράς συγκεκριμένων ενεργειών. Πριν από μερικά χρόνια το ενωσιακό εμπορικό επιμελητήριο είπε ότι θα αποσύρει την δραστηριότητά του αν αυξηθεί ε, ο ελάχιστος μισθός. Συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε για το ISTS Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα οι χώρες αυτές για περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς λόγους να επιβάλλουν περιορισμούς. Για το σημείο 9 τώρα, απελευθέρωση των δημοσίων προμηθειών. Είναι πιθανό ότι κάτι τέτοιο θα επιδίνωνε τις δημόσιες ε, υπηρεσίες στο Βιετνάμ, δηλαδή τις βασικές υπηρεσίες. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε πού ακριβώς θα περιληφθεί κάτι τέτοιο. Εφόσον υπάρχουν ήδη χαμηλά επίπεδα ε, ρυθμιστικών διατάξεων, εάν υπάρξει απελευθέρωση, οπωσδήποτε θα υπάρξουν περαιτέρω απολύσεις. Και για το σημείο 7, για την απελευθέρωση των ε, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και εδώ χαμηλά επίπεδα ρύθμισης και επίβλεψης και παρόλα αυτά επιδιώκεται περαιτέρω απελευθέρωση. Περαιτέρω μείωση ε, των ρυθμίσεων αυτό θα είναι ιδιαίτερα επιζήμιο και ενδεχομένως και αποσταθεροποιητικό για την οικονομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σειρά έχει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.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 Αλλάξτε καλύτερα μικρόφωνο γιατί μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Okay, new try. Thank you very much. Ωραία, ξαναπροσπαθώ λοιπόν. Ε, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω και να ζητήσω συγγνώμη και από το Διευθυντή των Επικεφάλων των Διαπραγματεύσεων ε, που δυστυχώς ε, ε, είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις, έπρεπε να παραστεί σε μια άλλη διαπραγμάτευση. Έχουν αναπληρώτρια. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των διαπραγματεύσεων μέχρι στιγμής, για να ανακεφαλαιώσω, ο έκτος γύρος έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα, πήγε καλά η πλευρά του Βιετνάμ ε, επιβεβαίωσε ότι ενδιαφέρεται να έχουμε ολοκληρώσει εντός του τρέχοντος τους ε, και θέλουν να διαπραγματευθούν στις διάφορες ομάδες εργασίας. Εμείς ε, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε στο τεχνικό επίπεδο τρία, επί τρία κεφάλαια, την κατάσταση των εμπορικών φραγμών, ανταγωνισμό μεταξύ άλλων. Επίσης σε κάποια άρθρα άλλων κεφαλαίων έχουμε σημειώσει πρόοδο. Συνολικά. Έχουμε κάνει ανταλλαγή σε μια δοσμολογική προσφορά. Ξέρετε ότι έχουμε πολλές, πολλά αιτήματα από την ευρωπαϊκή πλευρά να καλύψουμε πνευματικά δικαιώματα, δημόσιες συμβάσεις, κανόνες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λίγα μόνο σας αναφέρω. Commitment of Vietnam to engage also on these other sectors. Έχουμε μείνει λίγο πίσω λοιπόν στο τομέα των δασμολικών προσφορών στα tariff offers. Στόχος μας είναι να έχουμε ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα θετικό σε όλους τους τομείς. Για να σας τονίσω λίγο από τους ε, τομείς. που αναφέρθηκαν και στο ψήφισμα και από τους ομιλητές σε ό,τι αφορά τα φυτογειονομικά και υγειονομικά μέτρα Αυτό που θέλουμε είναι επιτόπου να έχουμε διαφάσεις για τους ε, εξαγωγείς. Έχουμε τη συμφωνία του ΠΟΕ, αλλά θέλουμε να διευκρινιστούν οι διατάξεις αυτής της συμφωνίας ώστε να διευκολύνονται οι εξαγωγεί ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να παραμένουν οι απαραίτητοι και δύο πλευρές έλεγχοι. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, καλή μεταχείριση των ζώων, το θέμα το διαπραγματεύεται η ομάδα του SPS των ε, υγειονομικών αυτογενομικών ε, διατάξεων. Το που θα μπουν όμω, αν θα μπουν στο κεφάλαιο τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν το λένε ξεκάθαρα για να αυτό. Σχολιάζουν ε, λέγοντα ότι δεν ξέρουν ακριβώ πού να ενταχθεί αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει δηλαδή εκεί κάποιο υπουργείο που να είναι αρμόδιο άμεσα για το θέμα αυτό τη καλή μεταχείριση των ζώων. Υπάρχουν επίση κάποια άλλα ε, στοιχεία τη βιώσιμη ανάπτυξη που σχετίζονται συγκεκριμένα με το, εμπόριο, το παράνομο εμπόριο ε, άγρια πανίδα. Οι Βιετναμέζοι όμως έχουν ε, ενδιαφέρον και συμφέρον να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Δεν έχουμε ακόμη όμως φτάσει ε, στο τελικό στάδιο. Στον τελευταίο γύρο σημειώσαμε σημαντική πρόοδο, είναι καλές οι συνομιλίες, αλλά εξακολουθούν να, να υπάρχουν ζητήματα από των οποίων δεν έχουμε ακόμη καταλήξει σε συμφωνία. Όπω και τα εργασιακά δικαιώματα, ένα θέμα που αναφέρθηκε. Βέβαια είναι μεγάλη προτεραιότητα της πλευράς της δικής μας να έχουμε ισχυρέ διατάξει στο κεφάλαιο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα δούμε λοιπόν πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε στον επόμενο γύρο. Τα σχόλια για τη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων τώρα. Το έχουμε ξαναπεί ότι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προτεραιότητα βασική. Το γνωρίζουν και οι Βιετναμέζοι. Θα θυμάστε ότι είχαμε διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Συμφωνία Συνεργασίας που έχουμε ήδη συνάψει με το Βιετνάμ. Ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα που διεξάγουμε με το Βιετνάμ ήδη είχε αρχίσει να ενισχύεται στο πλαίσιο του διμερούς διαλόγου. Έχουν γίνει δηλαδή πρώτες σχετικές συναντήσεις. Βέβαια και στη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου και σε όλες τις νέες συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου που συνάπτει η Κομισιόν προσπαθούμε να συσχετίσουμε αυτή τη ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συμφωνίες και την εφαρμοστικό τους ε, μηχανισμό σε άλλους τομείς τώρα, θα πρέπει να σας πω ότι το Βιετνάμ ε, είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο ότι αφορά όχι μόνο ε, την ολοκλήρωση, αλλά και την ε, κατάργηση των δασμών. Θέλουν να είναι ευρεία αυτή η κατάργηση των δασμών. Δεν έχουν ευθύς εξ αρχής αποκλείσει κάτι. Βέβαια, θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρξουν ε, μεταβατικές περίοδοι, αλλά δεσμεύονται να έχουμε μηδενικούς δασμούς μέσα στο χρονοδιάγραμμα που ορίζει το διαρμητικό έγγραφο που είχε συμφωνηθεί πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Παίρνω σε έναν άλλο τομέα που νομίζω ότι θα είναι και αυτός ενδιαφέρον για τα παραρτήματα του NTB. Θέλουμε να τηρηθούν τα διεθνή πρότυπα, να διευκολυνθεί το εμπόριο. Ήταν ανοιχτή η Βιετναμέζη σε ό,τι αφορά τα παραρτήματα για τους μη φραγμούς NTB. Υπάρχει σχετικός κανονισμός. Επίσης καλή ήταν η συζήτηση για τα πράσινα αγαθά και για τους δασμού που σχετίζονται με περιβαλλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες, το κεφάλαιο των υπηρεσιών. Και εκεί βλέπουμε να υπάρχει θετική δέσμευση από πλευρά Βιετνάμ. Διαπραγματευόμαστε επίσης το παράρτημα για την αυτοκίνητο μηχανία και τους σειρμούς πάλι στο παράρτημα των μετασμολογικών φραγμών. Θέλουμε να χρησιμοποιηθούν τα διεθνή πρότυπα και βλέπουμε να υπάρχει σχετική δέσμευση. Θέλουμε επίσης απλούστευση, διευκόλυνση του εμπορίου. Υπάρχουν αιτήματα και από τις δύο πλευρέ. Το σκέλος του ανταγωνισμού ε, το έχουμε ολοκληρώσει σε τεχνικό επίπεδο για το 20 Trust, τις ε, κρατικές επιχειρήσεις. Σε επίπεδο επικεφαλής διαπραγματεύσεων έχουμε καλές συζητήσεις και στο ψήφισμα αναφέρεται ότι ο κρατικός τομέας στο 40% της ε, οικονομίας του Βιετνάμ. Στόχος μας εδώ είναι να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε την ανταγωνιστική συμπεριφορά των κρατικών επιχειρήσεων στην αγορά του Βιετνάμ. Είναι ένα λεπτό ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχουν διάφορα συμφέροντα ε, στο όλο σύστημα του Βιετνάμ. Πάντως οι είναι καλές και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας σε αυτό το κεφάλαιο. Ένα τελευταίο σημείο. για τις δημόσιες προμήθειες, τους διαγωνισμούς. Πολύπλοκος τομέας, ιδίως ε, σε επίπεδο διαπραγματεύσεων με το Βιετνάμ. Δεν έχουμε προχωρήσει πολύ στις συζητήσεις για τους διαγωνισμούς. Έχουμε να καλύψουμε μεγάλο έδαφος ό,τι αφορά τα κείμενα που έχουμε μπροστά μας. Δεν έχω να σα δώσω συγκεκριμένη ενημέρωση για το που βρισκόμαστε. Δεν μπορώ να πίσω το έτοιμά σα σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο αυτών των δημοσιοπρομηθείων, διότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το στάδιο. Ακόμη και αν υπήρξε μια ανταλλαγή προσφορών. Για τα πνευματικά δικαιώματα για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Έχουμε κάνει προτάσεις, ε, εξετάζουν τις προτάσεις αυτές οι Βιετναμέζοι. Είναι... Καλές ε, οι συζητήσεις μας συνεχίζονται μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ. Πριν επανέλθουμε στον εισηγητή μας, ο Ντέβιντ Μάρτιν έχει ένα αίτημα. Παρακαλώ. Ε, δεν χρειάζεται να μιλήσω ακουστικά αυτά που θέλω να πω από άλλου. Κάποια σχόλια ο εισηγητή. Κύριε εισηγητά, έχετε κάτι να πείτε. Κύριε εισηγητά λέω. Σχόλια. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδης ηγητές για τις φιλικές και ανοιχτές παρατηρήσεις τους. Με χαρά βλέπω ότι το βασικό το περιεχόμενο κατά βάση του σχεδίου ψηφίσματος είναι αποδεκτό από όλες τις μεγάλες ομάδες. Ίσως θα πρέπει να χτενίσουμε κάποιες ε, λεπτομέρειες μέσω περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Ελπίζω ότι θα κλείσουμε πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι λεπτομέρειες μένουν, δεν θα υπάρχουν ουσιαστικές νέες αλλαγές. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε σύντομα λοιπόν το πακέτο και με χαρά να το υποβάλλω στην Επιτροπή έγκαιρα για να ψηφίσουμε όπως προβλέπετε τον Μάρτιο στην Ολομέλη. Ευχαριστώ. Ωραία. Προθεσμία τροπολογιών 27 Ιανουαρίου, 12 η ώρα το μεσημέρι. Θα ψηφιστεί στην επόμενη συνάντησή μας, 12-13 Φεβρουαρίου. Προχωρούμε στις ψηφοφορίες, ετοιμαστείτε. Σεβέρ. What problem?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 Let's Συμφωνήσαμε το σημείο 11 να ψηφιστεί τελευταίο. Προχωρούμε λοιπόν στο σημείο 12. Κοινωτι... Προσαρμογή του κανονισμού κοινοτικών στατιστικών για το εξωτερικό εμπόριο. Τροπολογία 7 υπέρ. Η ομάδα μου έχει δύο ερωτήσεις, πρόεδρε, συγγνώμη που το λέω τώρα. Θέλουμε να αλλάξουμε τον κατάλογο ψηφοφορίας για την τοπολογία 7 πίσω, ε, πλην το 10 το ίδιο και στο τέλος έχουμε επιφύλαξη. Εύκολα θα λυθεί, αλλά πρέπει να σας πω ότι στην τελική ψηφοφορία μπορεί να καταψηφίσουμε το κείμενο. Ε, απλά να σας ενημερώσω. Ωραία, έγινε η ανακοίνωση. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Το υπολογείο 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Το υπολογείο 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Το υπολογείο 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 1 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 12 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Αιτιολογικές σκέψεις, τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 4 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 5 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 6 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία για την πρώτη σε επιτοπίση όπως τοποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία. Ένας από το ΕΡΚ παραπάνω, εντάξει τώρα, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, ψηφίζουμε. Πέραση ψηφοφορία, Το ίδιο αποτέλεσμα. Ξέχασα να σα πω το αποτέλεσμα, αλλά είναι ίδιο. 19 υπέρ, 10 κατά. Σημείο 12. Σχέδιο σύσταση, διαδικασία σύμφωνη δρόμη για μια διεθνή συμφωνία. επιβολή δασική Νομοθεσία στη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφωνία με την Ινδονησία. Ε, σύμφωνη γνώμη είναι. Ναι, όχι, λέμε. Ονομαστικά. Ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Ομοφωνία 29 ψήφοι υπέρ. Συγχαρητήρια. τον Γιάννη Ξάντος. Σχέδιο ψηφίσματος για το ίδιο θέμα. Ίδιος εισηγητής. Συμβαστική τροπολογία 1. Μιλάμε για το σημείο 14 στην ημερήσια διάταξη. Υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Προφορική τροπολογία με αριθμό 1, αντιρρήσεις για να περάσει, για να δεχθούμε την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή. 9. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 6, συμβιβαστική 6 υπέρ, 6 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά αποχές απο, απορρίπτεται. Έλεγχος για την τροπολογία 18. Ηλεκτρονικός έλεγχος, την ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. συμβιβαστική 9 αποχές, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 11 συμβαστική υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προφορική τροπολογία 2. Οι για να δεχθούμε στην ψηφοφορία αυτήν. Όχι. Ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. 24 λέει ο πρόεδρος, αλλά για την 34 μιλά. 34 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 34 διορθώνει ο πρόεδρος. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 35 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 36 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή τελική ψηφοφορία άχετη ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας. «27 υπέρ, 2 αποχές, καμία ψήφος κατά συγχαρητήρια» προς τον εισηγητή. Θέμα 15. σχέδιο σύστασης για την ε, σύμφωνη γνώμη στην συνθήκη για τον πόδιο όπλων. Όχι ακριβώς δηλαδή, να επιτρέψουμε σε κράτη-μέλη να επικυρώσουν ε, τη σύμβαση αυτή εξ ονόματος της Ένωσης. Είναι συνθήκη, σύμβαση του ΟΗΕ που και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέλος του ΟΗΕ βεβαίως. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ψηφίζουμε ναι, όχι. Πέρασε. Ομοφωνία. Μπράβο κύριε Μάρτιν. Για το ίδιο θέμα, σχέδιο ψηφίσματος για την εφαρμογή της συνθήκης Εμπόδιο όπλων. Όπως ε, ξέρετε συμφωνήσαμε να υπάρξει ένα κοινό ψήφισμα με την ΑΦΕΤ. Οι τροπολογίες μας θα συμπεριληφθούν στο κοινό ψήφισμα. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμφωνία ε, τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή, δεκτή, 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Για την 11 θα κάνουμε έλεγχο, άρχεται η ψηφοφορία. 12, όχι 11. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρασε. Τροπολογία 13. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 14. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 15. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έλεγχος για την τοπολογία 18 Άρχιε την ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Τοπολογία 19. Υπέρ κατά αποχές Έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τοπολογία 19. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τελική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Ομόφωνα συγχαίρουμε τον εισηγητή. Item 17. 17. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία έρχεται. Πέρας. 27 υπέρ, 2 αποχές. 18 σχέδιο γνωμοδότησης για την πρόληψη και διαχείριση της αγωγής και εξάπλωσης χώρο κατακτητικών ξένων ειδών. Η συγγήτρια η Κάθριν Μπίεζα. Ας ψηφίσουμε λοιπόν. Τροπολογία 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις να ψηφιστεί θα γίνει κατά τμήματα ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. «28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται». 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 8 υπέρ,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 Λοιπόν, ήταν η 16 αυτή. Τώρα έχουμε την τροπολογία 2 κατά τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές. Λοιπόν, ας ελέγξουμε γιατί δεν είναι σαφές. Άρχεται το δεύτερο τμήμα. Πέρας. εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική, ωραία, ας ψηφίσουμε. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία άρχεται πέρας εγκρίνεται 27 ε, υπέρ ε, μία ψήφος κατά δύο αποχές 19. Γνωμοδότηση για τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Κορέας. Μία μόνο ψηφοφορία. Ονομαστική και άρχεται. Πέρας. 26 υπέρ, <clears throat> τρεις αποχές. Καμία ψήφος κατά. Συγχαίρουμε τον εισηγητή. 20. Αντίπεινα μέτρα της Κίνας κατά των εισαγωγών ίνου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει προφορική τροπολογία, έχει, υπάρχει καμία αντίρρηση. Όχι, ωραία, ας ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ονομαστική. Πέρας. 27 υπέρ, 0 κατά 2 αποχές. Συγχαίρουμε τον εισηγητή. Α, σε ποιον, δεν υπάρχει κανείς εισηγητής, ωραία, δεν συγχαίρουμε κανέναν. 21. Η, αυτή είναι η έγκριση των αποτελεσμάτων του τριμερού διαλόγου για τη διπλή χρήση. Η συγκητής μας είναι ο κύριος Φιέλνερ, προφορική ψηφοφορία για το αν θα επικυρώσουμε τη συμφωνία μας με το Συμβούλιο, Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρα Λοιπόν, 25 υπέρ, 0 κατά 4 αποχές, συγχαίρουμε τον εισηγητή μας ο οποίος ε, έκανε εξαιρετική δουλειά, ε, ήμουν παρόν και το διεπίστωσα. Το... Ας περάσουμε τώρα, επανερχόμενοι, στο πρώτο θέμα της ψηφοφορίας. Ένα θέμα που θα μας απασχολήσει κατά πολύ είναι εισηγητής ο κύριος Κρίστοφερ Φιέλνερ και αφορά τον κανονισμό ε, εισαγωγών dumping. Θέλετε να πείτε τίποτα? Ευχαριστώ για τη στήριξή σας, ε, για την διπλή χρήση. Ήταν πολλή δουλειά και τα πήγαμε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την εργασία που έγινε για το μηχανισμό ε, για το εμπόριο ε, και την άμυνα. Για το μέσο εμπορικής άμυνας, συγγνώμη, θα πρέπει να θυμάστε ότι αρχίσαμε τον περασμένο Ιούνιο-Ιούλιο την εργασία μας. Σε πέντε μήνες λοιπόν καταλήξαμε παρά τις διακοπές. Θα πρέπει ίσως να μπούμε στο βιβλίο Γκίνες για το θέμα αυτό. Ήταν το πιο ε, επίμαχο τμήμα της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης και νομίζω ότι επιτύχαμε σχεδόν όλους μας τους στόχους γιατί αν εξετάσετε το κείμενο υπάρχουν πολλές γκρίζες περιοχές δηλαδή 11 συμβιβασμοί που καλύπτουν σχεδόν όλες τις ε, σημαντικές πλευρές του θέματος. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια εξυγχρονισμού του μέσου εμπορικής άμυνας, του μηχανισμού εμπορικής άμυνας. Είπα λοιπόν ότι τα καταφέραμε σχεδόν παντού, διότι σε δύο από τους 13 τομείς δεν επιτύχαμε ε, συμβασμούς. Φυσικά είναι οι πιο επίμαχη τομείς. Και θα ψηφίσουμε λοιπόν γι' αυτό. Ε, υπάρχει αλληλεξάρτηση για πολλούς συναδέλφους αυτών των δύο τομέων. Θα προτιμούσα να αναβληθεί η ψηφοφορία, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό, γιατί το βασικό είναι να περάσει το μήνυμα στην Κομισιόν ότι η υποβολή τόσο περίπλοκων θεμάτων στο τέλος της θητείας δεν μας βοηθάει. Παρακαλώ λοιπόν συνάδελφοι, από σήμερα μέχρι την Ολομέλεια να ε, πάρουμε το χρόνο για να διαπραγματευτούμε για να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις για αυτά τα δύο σημαντικά θέματα. Γιατί αν το επιτύχουμε θα ψηφίσουν μαζί ε, οι ομάδες και θα είναι σαφέστερες και οι διαπραγματεύσεις με το Συμβουλίο. Γιατί ελπίζω να αξιοποιήσουμε αυτές τις δύο εβδομάδες. Ευχαριστώ ωστόσο όλους όσους συμμετείχαν. Νομίζω ότι είναι θαυμάσιο το αποτέλεσμα αυτών των 11 συμβασμών και θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτά που επιτύχαμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να ψηφίσουμε. Έχω ένα σημείο από τη γραμματεία που μας λέει ότι οι τροπολογίες 216 και 325 αντίθετα με ό,τι αναφέρεται στην ε, λίστα ψηφοφορίας δεν έχουν αποσυρθεί. Θα τις θέσουμε σε ψηφοφορία. 216-325. Αυτές οι δύο τροπολογίες θα τεθούν σε ψηφοφορία, διότι δεν έχουν αποσυρθεί. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αχ, με συγχωρείτε. Λάθος έκθεση. Λάθος έκθεση. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πολύ μ' αρέσει να βλέπω έτσι, πολύ γκρίζο. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δέσμη 1. Τροπολογίες 1 έως 7 και άλλες τροπολογίες. Δέσμη 1 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνονται, τροπολογίες αυτές. Δες τροπολογιών 2, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και δέσμη 2. Τρίτη δέσμη τροπολογιών, υπέρ, κατά, αποχές να ελέγξουμε, δεν είμαι βέβαιος για το αποτέλεσμα. Δέσμη τροπολογιών υπαριθμών 3, άρχεται η ψηφοφορία. Έληξη ψηφοφορία. Εγκρίνονται οι τροπολογίες αυτές. Δέσμη 4, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Όχι 13. Υπέρ. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι, δεν συμφωνείτε. Να ελέγξουμε την τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τώρα που πηγαίνουμε. Τροπολογίες 197-199. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνονται. Δέσμη 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δέσμη 6. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είμαι βέβαιος, να ελέγξουμε για τη θέσμη τροπολογιών παριθμών 6, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα περνάμε στην τροπολογία απορρίφθηκε. η δέσμη 6. Συγγνώμη, νόμιζα ότι το είχα, το είχα πει. Τώρα περνάμε στην τροπολογία 160 σε τρία τμήματα ή μάλλον πέντε τμήματα. Πρώτο τμήμα Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε το τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μπορούμε παρακαλώ να ελέγξουμε το δεύτερο με κασπάρι; Ποιο λέτε? Το δεύτερο. Το δεύτερο τμήμα. Ας ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 160. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τι γίνεται τώρα με την 7η δέσμη τροπολογιών. Καταπίπτει. Μάλιστα, καταπίπτει. Το ίδιο συμβαίνει και με, την τροπολογία 154 ή μάλλον και 156. 178. 158. Όχι. Ψηφίζουμε την 158. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. 158. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε 91 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 91 άρχη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 92. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87. Τι γίνεται. Καταπίπτει. Όχι. Ψηφίζουμε το 87 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 151 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 89 και 90 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε τις 89 και 90 άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 185. Πέντε τμήματα. Πρώτο τμήμα της τροπολογίας 185 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα ψηφιπέρ, Κατά αποχές εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα ψηφιπέρ, Κατά αποχές εγκρίνεται. 179 καταπίπτει. Μάλιστα. Όπως και η 181. 182, 183, 184. Πάμε στη δέσμη τροπολογιών παριθμών 8. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπέρθμο 10, ψήφι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Δέσμη τροπολογία υπέρθμο 9, ψήφι υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 297 ψήφι υπέρ. Δεν έχει καταπέσει ψήφι υπέρ της 297. Κατά αποχές απορρίπτεται. Όχι, συγγνώμη. Έχετε δίκιο. Είχαμε και τη 291 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε τη 291. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29. κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ελέγχουμε την 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 309 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93, 93 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Η 93 θέλετε τι, να ελέγξουμε. Εντάξει. Ελέγχουμε την 93. Έληξε ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 95. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 102 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, όχι, να ελέγξουμε. 102. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 111. Ψήφι υπέρ. 111. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11. Ψήφι υπέρ. Τι να ελέγξουμε. Την 111. Να ελέγξουμε την 111. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Compromise Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 165. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτεται 188. 189 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 196 η δεκτονική ψηφοφορία και έλεγχος για την 189 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 206 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται.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 206. Δεν έχει αποσυρθεί, την ψηφίζουμε. 216 υπέρ κατά εποχές δεκτή. at ε, and now let's move to 226. 226. υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 228 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 232 και 233 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 234 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 286 υπέρ κατά δεκτή. 287 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 287. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 311 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 216. Έλεγχος για την 311. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 216 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το 225. Κακώς αναφέρεται ότι είχε αποσυρθεί. Δεν είχε αποσυρθεί. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 325. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 339. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1 υπέρ καταπίπτει. Καταπίπτει. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, διορθώνει ο πρόεδρος. Αιτιολογική σκέψη 4. Οι τροπολογίες είναι οι 40 και 41. Υπέρ των 40-41 κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 46 είναι ίδια με τη 42. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ Ξέρω ότι είναι κάπως ε, Προβληματικό ο κατάλογο τη γιατί γίνανε αλλαγέ, αλλά κάτι δεν πάει σωστά στη 44. 44 λέει ότι καταπίπτει αν εγκριθεί η τροπολογία 44. Άρα μάλλον δεν τραβάει, δεν υπάρχει διέξοδο. Μπορείτε να μα πείτε τι ακριβώ συμβαίνει με την τροπολογία 44 και τη 43. Η 43 τι έγινε, κατέπεσε. Η 43 καταπίπτει, η 44 ψηφίζεται. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές. Θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για τη 49. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 50. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τι έγινε, τι κατέπεσε εδώ. 57. Υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τοπολογία 57. Πέρας της ψηφοφορίας. Απολύπτεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 58 κατέπεσε ήδη. Όχι. Δεν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. οι τροπολογίες 59 και επέκεινα κατέπεσαν. Ναι. Και το ίδιο ισχύει με την 337. Όχι, δεν κατέπεσε. Ψηφίζουμε την 337. Υπέρ. Κατά. Λοποχές. Τι, τι ψήφισε η δεν το κατάλαβα. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 337 τις ψηφοφορίας. Δεκτή. Η 65 κατέπεσε. ...231 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 66 και 67 και 68 και 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Η 70 κατέπεσε. Η 88 υπέρ κατά εποχές δεκτή. 72 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έλεγχος για την 72. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 230 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Ε, απορρίπτεται, συγγνώμη. 80 και 81 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 82 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται, απορρίπτεται. Και η τελική ψηφοφορία. Αρχίζουμε. Είναι, ψηφίζουμε την πρώτη της Επιτροπής όπως τοποποιήθηκε καταρχάς. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Γκρίνεται 24 ψήφοι υπέρ, 6 κατά, 0 αποχές. Να ψηφίσουμε τώρα το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται. Πέρας. ίδιο συσχετισμό 24 υπέρ κατά 0 απόχέ. συγχαίρουμε τον εισηγητή Τι προτείνετε κύριε εισηγητά για τα επόμενα βήματα Θέλουμε να υποβληθεί στην Ολομέλεια το ταχύτερο για να έχουμε έτσι ε, ισχυρότερη θέση για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Πρόεδρος, ωραία. Για να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις πρέπει να εγκρίνουμε την εξή απόφαση να... <coughs> να εγκρίνουμε... Όχι, όχι, ο Όχι, δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε τώρα τις διαπραγματεύσεις. Όχι, δεν θέλουμε διαπραγματεύσεις πριν την Ολομέλεια. Γιατί όπως όλοι ξέρετε Υπάρχουν πολλοί ε, που δεν είναι παρόντες εδώ αυτή τη στιγμή που έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις. Θα πρέπει λοιπόν να περάσει στην Ολομέλεια το θέμα αυτό. Ωραία. Λίγη η ώρα ψηφοφοριών. Ευχαριστώ πολύ. 22. Εκεί. Thank you. Παρακαλώ όσοι βγαίνουν ε, να συντομεύσουν και να βγουν χωρίς πολύ φασαρία.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 Okay. So Delegation to India is item 24. Yes. Ah, it's next. Okay, okay, okay. So it is right now? Yeah, no, now we have 22. No, only two items. They are very brief. Okay. okay. Sorry. No, no problem. Okay. Shall we move on? Λοιπόν, συνεχίζουμε. 22. Μακροοικονομική βοήθεια στην Τινησία. Η, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση να δώσουμε οικονομική βοήθεια στην Τινησία. Δεν είναι δυσχερές το θέμα. Έχει εγκριθεί η συμφωνία πλαίσιο με το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Πρέπει λοιπόν να εγκρίνουμε τι μορφή. Το ποσό θα το αποφασίσει η Επιτροπή. Είμαι εισηγητής. Έχω υποβάλει λίγες τροπολογίες ε, για να συμμορφωθεί η ορολογία με την ορολογία του, της Συμφωνίας Πλαισίου. Ωστόσο, μεταξύ, το Συμβούλιο μου είπε ότι θα πρέπει να αυξηθεί το ποσό. Τους απήντησα ότι το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να δεχθεί αυτή την αύξηση μόνο εάν εγκριθεί κατά την τρέχουσα θητεία το θέμα αυτό. Να μην υπάρξει κίνδυνος να ε, μην προλάβουμε. Το συζήτησα και με τις πολιτικές ομάδες που συμφωνούν με την ίδια προϋπόθεση. Και με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. η οποία ήταν πολύ ανοιχτή να συντάξουμε δηλαδή μια γνωμοδότηση που να μην αναφέρει το ποσό. Συμφώνησα τα εξή με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Λοιπόν, θα υποβάλουν το αργότερο σήμερα γραπτός αίτημα στα άλλα δύο θεσμικά όργανα για αύξηση του ποσού. Θα λάβουμε τη γνώμη της Επιτροπής Προϋπολογισμών που θα δεχθεί. Θα υποβάλω ε, την τροπολογία εγώ ο ίδιος και θα εγκριθεί πριν το τέλος της θητείας. Καλή απόφαση είναι αυτή νομίζω. Δεν κινδυνεύει ο βασικός μας στόχος και εφόσον συμφωνούν ε, να υπάρξει αύξηση τα άλλα δύο ε, θεσμικά όργανα δεν θα έπρεπε να το αρνηθούμε. Δεν μου έχει ακόμη σταλεί το γραπτό αίτημα. Θα περιμένω μέχρι σήμερα το βράδυ. Λοιπόν, συζήτηση. Σκιώδης του ΕΛΚ Νόρα Μπέρα. Παρακαλώ. Βεβαίως, σας βλέπω. Παρακαλώ. Είμαι μείωψα, αλλά όχι και τόσο. Ε, κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει επίγοντα προβλήματα της τυνησίας, αλλά ε, ανταποκρίνεται και στην, ανάγκε στις ανάγκες της πολιτικής και δημοκρατικής. Ξέρετε ότι υπάρχει βαθιά μεταρρύθμιση εδώ και τρία χρόνια χάρη στο θάρρος και τον αλτρουισμό των πολιτών. Είμαστε τώρα σε νέα φάση αυτή τη διαδικασία αλλαγή ε, πρόσφατα. Είχαμε δύο μεγάλε δημοκρατικέ κατακτήσει που επικυρώθηκαν από τη νέα συντακτική συνέλευση. Άκουσα επίση να αναγνωρίζεται συνταγματικά η ισοτιμία όλων των πολιτών και ανδρών γυναικών έναντι του νόμου χωρί καμία διάκριση. Αυτό είναι πρώτη φορά που συμβαίνει στον αραβικό κόσμο και θέλω να το χαιρετήσω. Επίσης αναγνωρίζεται η ελευθερία συνείδησης και η θρησκευτική ελευθερία. Έτσι λοιπόν η Τινησία απορρίπτει τελειωτικά την Σαρία. Έτσι λοιπόν η Τινησία προχωράει προς την κατεύθυνση ε, οικοδόμησης ενός δημοκρατικού κράτους, ενός κράτους δικαίου, αλλά ξέρουμε ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί σε συνθήκες οικονομικής ε, κρίσης ε, και αυτό μπορεί να προκαλέσει ε, επιστροφή στην πολιτική αστάθεια και τη βία. Θα πρέπει λοιπόν να συμβάλλουμε ούτως ώστε να κατοχυρωθούν τα δημοκρατικά κεκτημένα επειδή έχουμε προνομιακές σχέσεις με την Τινησία και με βάση τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε τον Νοέμβριο του 2012 κατά συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Τινησία πρέπει να στηρίξουμε αυτήν την δημοκρατική μετάβαση. Πρέπει να ελπίσουμε ότι η Ισία σταδιακά θα μπορούσε να ενταχθεί στην ε, εσωτερική μας αγορά και γι' αυτό θα πρέπει ανεπιφύλακτα να ε, είμαστε υπέρ μιας μακροοικονομικής βοήθειας που θα επιτρέψει την Ισία να χρηματοδοτήσει τις πολιτικές της. Χαιρετίζω την πρότασή σας κύριε Πρόεδρε που προτείνει την αποδοχή της αύξησης του ποσού της βοήθειας και θα παρακολουθήσουμε προσεκτικά το πώς θα δεσμευτούν το Συμβούλιο και η Επιτροπή για να ικανοποιήσουν αυτό το αίτημα. Τι μορφή τώρα θα έχει αυτή η βοήθεια. Η Κομισιόν μας προτείνει μια βοήθεια που θα είναι αποκλειστικά μέσω δανείων. Κάτι που είναι σύμφωνο με τον κανόνα της ε, διοργανικής συμφωνίας. Θα μπορούσε η Κομισιόν να δώσει και βοήθεια μέσω χορηγιών με βάση την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και του μέσου εισοδήματος των κατοίκων της. Ε, έχει γίνει κάτι παρόμοιο σε προηγούμενες περιπτώσεις, για παράδειγμα στη Γεωργία. Τους δώσαμε 50% ε, της βοήθειας ως χορηγία. Και επειδή το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης των δύο χωρών είναι συγκρίσιμο, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να προτείνουμε και τέτοιου τύπου βοήθεια προς την Τινησία. Ευχαριστώ πολύ και χαιρετίζω την προσπάθειά σας ε, μέσω της τροπολογίας που υποβάλλετε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Άλτερ. Καζάκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εισηγήτριά μας, η σκιώδη δεν είναι εδώ. Να σας παρουσιάσω εν συντομία τη θέση μας. Αυτή η συμφωνία που έχουμε με την Τινησία μας ε, χορηγεί ε, αμοιβαία ωφέλη και βοηθάμε την, οικονομική την πολιτική μετάβαση και την οικονομική ανάπτυξη της Τινησίας και θα θέλουμε να υποστηρίξουμε περαιτέρω τους πολιτικούς κοινωνικούς συγγνώμη, τις πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται και επειδή είναι πολύ ευαίσθητη η οικονομική κατάσταση της χώρας η προστιθέμενη αξία της συμφωνίας αυτής θα είναι να βοηθήσει την Τινησία να δημιουργήσει ένα σταθερό μακροοικονομικό πλαίσιο προωθώντας και μια βιώσιμη, ένα βιώσιμο ισοζύγιο πληρωμών και ένα βιώσιμο δημοσιονομικό πλαίσιο όπως έχει συμφωνηθεί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η πολιτική και οικονομική στήριξη τη Ένωση προ την Ισία θα βοηθήσει επίση να ενισχυθεί η δέσμευση τη κυβέρνηση να κάνει μεταρρυθμίσει και η προσδοκία τη για στενότερε σχέσει με την Ένωση όπω ανέφερε και η συνάδελφο από το ΕΛΚ. Ευρύτερα το πρόγραμμα θα είναι θετικό μήνυμα και προς άλλες χώρες της περιοχής ότι η Ένωση είναι διατεθειμένη να στηρίξει εκείνους που ξεκινούν μια σαφή πορεία προς πολιτικές μεταρρυθμίσεις σε περιόδους οικονομικών δυσχεριών. Αυτό βεβαίως είναι τμήμα της πολιτικής της Ένωσης για το νότιο τμήμα της Μεσογείου και της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας για να έχουμε βιώσιμα αποτελέσματα και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις εξελίξεις επί τόπου στις χώρες αυτές, αν και μερικές φορές, αυτό ε, περιπλέκει την κατάσταση και μπορεί να μας φέρει ενώπιον απροσδοκήτων καταστάσεων. Θα πρέπει να διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο δέσμευση στις σχέσεις, στις σχέσεις μας με την Τινησία και γι' αυτό δεν θα πρέπει να υπάρξουν καθυστερήσεις στην εκταμείευση αυτής της ενίσχυσης. Γιατί θα ήταν αντίθετο αυτό προς τη δέσμευσή μας και τις προσπάθειές μας να βοηθήσουμε την Τινησία για πολιτική ανάπτυξη και οικονομική προσέγγιση. Υποστηρίζουμε λοιπόν την αύξηση του ποσού της μακροοικονομικής βοήθειας εφόσον δεν θα καθυστερήσει την εκταμίευση της βοήθειας αυτής. Ευχαριστώ. Επόμενος, συντηρητική, Ζάχραντιο. Δεν έχω να κάνω κάποια ουσιαστική ε, παρατήρηση κύριε Πρόεδρε. Ήμουν πολύ σύντομος. Σκά Κέλλερ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τους επένους ε, που ακούστηκαν για την Τινησία, τις ε, μεταρρυθμίσεις, την πρόοδο που έχει εκτελεστεί. Όμως, το θέμα είναι με αυτή τη βοήθεια εμείς πώς συνεισφέρουμε Καταρχήν δεν είμαστε αντίθετοι βέβαια, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε. Δηλαδή να μην οδηγήσουμε σε υπερχρέωση μια ακόμη χώρα που θα είναι πολύ δύσκολο μετά να βγει από αυτή την κατάσταση. Δίνουν μια γενική δημοσιονομική υποστήριξη με τη μορφή δανείου. Ξέρω πώς ε, γίνονται αυτά, αλλά θα συμβάλλει κάτι τέτοιο σε θετικές μεταρρυθμίσεις που βλέπουμε να γίνονται στην την Ισία. Μήπως να βρούμε μια άλλη μορφή και να μην δημιουργήσουμε ένα τεράστιο χρέος για την, ε, την Ισία. Το ποσό αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο για μια μικρή χώρα σαν την Ισία. Μιλάμε εδώ για ένα πολιτικό μήνυμα που θέλουμε να εκπέμψουμε. Μήπως αυτό θα μπορούσαμε να το εκπέμψουμε διαφορετικό τρόπο. Τι είδους μόχλευση έχουμε ώστε να πετύχουμε ε, την αξιοποίηση των κονδυλίων που θέλουμε να διαθέσουμε για να έχουμε πρόοδο επιτόπου. Καταρχήν λοιπόν δεν έχουμε αντιρρήσεις, αλλά πρέπει να είναι σαφής η στόχοι μας. Πρέπει να μην ε, προχωρήσουμε ε, ελαφρά την καρδία χωρίς να το σκεφτούμε το αποτέλεσμα που θα πετύχουμε. Πολ Μέρφυ από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ δεδομένου του ιστορικού ρόλου της Ευρώπης στην περιοχή, την ευρύτερη και στην Ισία ιδιαίτερα, που είχε στηρίξει δηλαδή τη δικτατορία του Μπεν για παράδειγμα, ε, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ε, στο πώς ε, παρεμβαίνουμε στην πολιτική, στην Τινησία και τι είδου συμφέροντα μπορεί να είναι από πίσω. Φυσικά δεν δίνουμε χρήματα γιατί ποτέ είναι σαφές ότι οι εκταμιεύσεις ε, θα ε, γίνονται μετά από θετική αξιολόγηση εκ μέρους του Ιθνούς Ταμείου και θα πρέπει βέβαια οι Κομισιόν την Ισία να συμφωνήσουν με ένα μνημόνιο συνεννόησης για συγκεκριμένες διαθροτικές μεταρρυθμίσεις. Μνημόνιο συνεννόησης λοιπόν μεταξύ την ΙΣΙΑ Κομισιόν. Αυτό όμως δεν υπάρχει. Εμείς δηλαδή ποτέ θα πρέπει να συμφωνήσουμε να δώσουμε χρήματα με κάποιες προϋποθέσεις που δεν τις βλέπουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση, δεν μπορούμε να κάνουμε ανάλυση ε, και είναι στο κάτι τέτοιο. Το πρόγραμμα όμως του Δημοσιονομικού Ταμείου είναι το αναμενόμενο. Μία νεοφιλελεύθερη συνταγή. Το αναμενόμενο. Δημοσιονομική εξυγίανση που σημαίνει αύξηση φόρων, κυρίως φόροι οι οποίοι σπράττονται από τον απλό κόσμο, τους εργαζομένους, τους ε, μικρούς αγρότες και όχι από τους πλούσιους οι επιδοτήσεις, αύξηση ίσως σε τιμές, ρεύματο ρεύματος, ενέργειας για εξοικονομήσεις πόρων. Όλα αυτά τα μέτρα από κοινού προκάλεσαν αντιδράσεις ε, στις αρχές Ιανουαρίου. Αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι χαιρέτησαν αυτές τις αλλαγές, αυτοί που έκαναν την επανάσταση στην Τινησία. Εγώ δεν είμαι υπέρ της χρήσης πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, προσθήκη ακόμη μεγαλύτερων, ε, περισσότερων μάλλον όρων σε ένα νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα. Εμάς μας ενδιαφέρει ο απλός κόσμος. Και σε ό,τι αφορά το χρέος, ε, η μόνη αναφορά ε, λέω ότι είναι βιώσιμο το χρέος, αλλά πριν από πάνω από ένα χρόνο στο Κοινοβουλή είχαμε πει ότι είναι παχθές το χρέος ε, αυτών των περιοχών στη Βόρεια Αφρική, ιδίω στην Τινησία, όλα αυτά προκλήθηκαν από τη δικτατορία, από το καθεστώς, όπως και σε άλλες χώρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, δεν είναι μη δημοκρατικό να μην έχουμε αυτό το μνημόνιο συνεννόησης πάνω στο οποίο βασίζεται η εκταμείευση των ε, πόρων και δεν ξέρουμε και πάνω σε ποιες βάσεις και τι θέλει να διαπραγματευτεί η Κομισιόν με την Τινησία. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Σα ακούσουμε τώρα την εκπρόσωπο της ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Ζάιντελ. Yes, thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, η κυρία Ζάιντελ δεν ήταν. Α, η κυρία Ζάιντελ είναι για το επόμενο θέμα. Ο κύριος Τέμπρα. Μόνο για τα πρακτικά είναι για να διορθώσουμε το όνομά σας. Καταρχάς να σημειώσω ότι η Επιτροπή υποστηρίζει βεβαίως τις τροπολογίες που προτείνει η συγγήτρια και που θα ευθυγραμμίσουν ακόμα περισσότερο το κείμενο. Με αυτό με τις επιχειρήσεις στην Κυργιζία και την Ιορδανία. Να αντιδράσω, να απαντήσω μάλλον στην ιδέα που πρότεινε το Συμβούλιο για την αύξηση στα 300 της βοήθειας. Κατά την άποψη της Επιτροπής αυτό θα αποτελέσει, περιλαμβάνει καλή αιτιολογία. Η οικονομική κατάσταση είναι κρίσιμη. Υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα τρέχουσων συναλλαγών και ε, δημοσιονομικό πολύ, χαμηλό, πολύ υψηλότερο από αυτό που προβλεπόταν στο πρόγραμμα του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου με μικρή ανάπτυξη, κάτι που θέτει ακόμα σε μεγαλύτερο κίνδυνο την ε, αλλαγή του καθεστώτος στην στιγμή που εμφανίζεται και που, ορί, που τοποθετείται στην κυβέρνηση μια τεχνοκρατική ομάδα που προσπαθεί να εφαρμόσει μια σειρά προγραμμάτων μεταξύ των οποίων και του ΤΑΦ. Πιστεύουμε ότι η αύξηση της βοήθειας αποτελέσει ένα καλό μήνυμα. Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις κατά την άποψη της Επιτροπής είναι περιορισμένες και διαχειρίσιμες. αυξηση 4-5 4,5 εκατομμυρίων ε, στον προϋπολογισμό της Ένωσης για τα επόμενα δύο χρόνια. Τέθηκε μία ερώτηση από την Γαλλίδα Ευρωβουλευτή που αφορούσε το ότι γιατί δεν χρησιμοποιούσαμε κάποια στοιχεία ενίσχυσης. Αυτό εξηγείται στην εξάντε αξιολόγηση. Δυστυχώς η Τινησία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να λάβει ενισχύσεις, ε, στοιχείο ενισχύσεων λόγω του σχετικά υψηλού ανα, ΑΕΠ ανακάτοικο. Ένα άλλο κριτήριο που χρησιμοποιούμε είναι το πώς ε, αντιμετωπίζουν οι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οργανισμοί μια χώρα. Ε, η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ δεν, δεν δίνουν πρόσβαση στην Ινησία σε οποιαδήποτε δημοσιονομικά εργαλεία που έχει που έχουν. Η προσέγγιση μας είναι λοιπόν συνεπής με την ε, ε, τάση μας να χρησιμοποιούμε δάνεια και όχι δωρεές, όλο ένα και περισσότερο. Ως προς τα άλλα σχόλια που τέθηκαν, το Μνημόνιο Συνεννοήσεως. Ένα σχόλιο που μόλις έγινε Βεβαίως υπάρχουν προϋποθέσεις και όροι, αλλά πρώτα πρέπει να έχουμε έγκριση των αποφάσεων από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πριν ξεκινήσουμε να διαπραγματευόμαστε και να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεννόησης δανείου. Προφανώς και θα υπάρξει ωστόσο. Αυτό είναι σύνηθις πρακτική. Αλλά θα, και η ενίσχυση θα ε, εξαρτηθεί από τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει το μνημόνιο. Τήρηση των προϋποθέσεων του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ και άλλες ε, υποχρεώσεις, φορολογική μεταρρύθμιση, ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής ασφάλειας για να καλυφθεί ε, το, για να μειωθούν οι επιπτώσεις τους πλέον ευάλωτους από τις αύξησεις των τιμών που θα απαιτηθούν για δημοσιονομικούς λόγους, καθώς και μέτρα εμπορίου και επενδύσεων που απαιτούνται για την κατασκευή, για την οικοδόμηση ισχυρότερων σχέσεων μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Τινησία. Σε ό,τι αφορά την, ε, το δημόσιο χρέος, είναι γεγονός ότι θα αυξηθεί το χρέος, αλλά το επίπεδο χρέους ε, τη Τινησία ε, είναι σχετικά διαχειρίσιμο. Από την άποψη αυτή λοιπόν, η πρόταση είναι εύλογη και διαχειρίσιμη. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ. Υπάρχει προφανώς υποστήριξη για την σύμφωνη γνώμη και όντως είναι μια πολύ επίκαιρη πρωτοβουλία. Προθεσμία για τις τροπολογίες, η άλλη πέμπτη μεσημέρι, 12 η ώρα. Το Συμβούλιο ζήτησε παράταση της προθεσμίας παρεπιπτόντος για το αίτημα να αυξηθεί το ποσό μέχρι αύριο. Αλλά το ίδιο θα ισχύσει και την Επιτροπή βεβαίω. Σημείο 23. συμφωνία μεταξύ Ένωση και μια σειρά χωρών Αυστραλία, Βαζιλία, Καναδά, Χονγκ Ινδία και Ιαπωνίας για τι τροποποιήσεις των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στους πίνακες της Βουλγαρίας και της Ρουμανία ως αποτέλεσμα της προσχωρησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από την συμφωνία GATS. Ο Γιάνν Ζάχαραντιλ είναι ο εισηγητής μας, στον οποίο δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τα είπατε όλα τα σημαντικά για το θέμα αυτό η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι μέλη, ήταν μέλη του ΠΟΕ πριν προσχωρήσουν στην Ένωση. Μετά χρειάστηκε να αλλάξουν τις ε, δεσμεύσεις του στον τομέα των υπηρεσιών, τροποποιώντας ε, τους πίνακες των ΓΚΑΤΣ, ούτω ώστε να υπαχθούν οι δεσμεύσεις της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη βάση του ΓΚΑΤΣ στους ε, περιορισμούς της Ένωσης για την αντιμετώπιση της πρόσβασης στην αγορά. Για τον λόγο αυτό, οι δύο αυτές χώρες θα πρέπει να προσφέρουν, να παρέχουν στις χώρες του ΠΟΕ την ίδια ε, αντιμετώπιση, ε, ιδίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, όπως και στα κράτη της Ένωσης. Η Βουλγαρία δε ιδιαίτερα θα πρέπει να επιτρέψει την ε, είσοδο δαπών εταιριών στον τομέα της ασφάλισης και η Ρουμανία ε, την είσοδο ασφαλιστικών υπηρεσιών στην δική της ε, χώρα. Εγώ προτείνω στην Επιτροπή μας να δοθεί η σύμφωνη γνώμη προς την συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ. Οι σκιώδεις εισηγητές, Πέτρε Στάσνη. Ευχαριστώ όπως αναφέρθηκε, τεχνικό θέμα, τεχνική σημαντική συμφωνία. Είναι παρόμοια με αυτή που είχε υπογραφεί το 2007 νομίζω όταν η Ένωση έγινε Ένωση των 25. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν κατέγραψαν τους περιορισμούς αυτούς και έχουν το δικαίωμα, είχαν το δικαίωμα να το κάνουν. Οχτώ χώρες ήταν αρχικά, πέραν αυτών ήταν και η Κίνα και το Μεξικό που αποσύρθηκαν κατόπιν και έμειναν οι χώρες που αναφέρονται τώρα. Έξι χώρες που υπέβαλαν ενστάσεις στον περιορισμό, στους περιορισμούς κάποιων σε κάποιους περιορισμούς της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Νομίζω ότι είναι σωστό, γι' αυτό και εγώ και η πολιτική μου ομάδα προτείνουμε να δοθεί συνένεση, σύμφωνη γνώμη στη σύμφωνη αυτή. Ο Μπερτ Λάγκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο, το άρθρο 21 Όντω, υποχρεώνει τα, κράτη, τα με κράτη στον ΓΑΤ να παρατείνουν τις διαπραγματεύσεις από τη στιγμή ωστόσο που υπάρχουν αλλαγές και η προσχώρηση των δύο χωρών Βουλγαρίας Ρουμανίας οδηγεί σε τέτοιες αλλαγές ζήτησαν παράταση έξι χρόνια, έξι χώρες. Στο αναμεταξύ συνήφθησαν, ολοκληρώθηκαν ε, οι διαπραγματεύσει όπως αναφέρθηκε στον τομέα της, ε, των ασφαλιστικών υπηρεσιών, άλλαξε η, άλλαξαν οι προθέσεις πρόσβασης στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Η λύση είναι θετική κατά την άποψή μας και εμείς συμφωνούμε με την πρόταση του εισηγητή. Θα θέλαμε να δοθεί η σύμφωνη γνώμη και για πολιτικούς λόγους βεβαίω, διότι εμείς τα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου σεβόμαστε τα μέτρα της διατάξεις του ΠΟΕ, θέλουμε πολυμερή αντιμετώπιση των διαφορών και αυτό ε, δείχνει ότι περνάμε ένα μήνυμα για ταχύ επίλυση τυχών διαφορών. Στο ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων για τις υπηρεσίες τέζα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να τιμήσουμε τις υποχρεώσεις μας έναντι του ΓΚΑΤ και να δίνουμε παράδειγμα. Ο σκιώδης ηγετής μας δυστυχώς είναι ε, στη Ρουμανία οπότε δεν μπορεί να είναι παρόν αλλά τα λέω εγώ. Κύριε Ζάιντελ από την Επιτροπή αυτή τη φορά. Ε, ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι εντελώ τεχνική είναι απόρρια της διαδικασίας ε, που πρέπει να εφαρμοστεί στον ΠΟ. Οι διαπραγματεύσεις έχουν κλείσει εδώ και μερικά χρόνια. Υπήρχε ένα διαδικαστικό πρόβλημα για την υπογραφή. Αλλά τώρα μπορούμε να υπογράψουμε αυτές τις συμφωνίες. Γι' αυτό ευχαριστούμε πολύ την ε, σύμφωνη γνώμη σας. Ο πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Ωραία, έχει τελικά σχόλιο εισηγητής. Όχι, λέει ο Ωραία, λέει ο πρόεδρος. Ε, προθεσμία η προσεχής Παρασκευή μεσημέρι για υποβολή τροπολογιών. Θα το εγκρίνουμε ως Επιτροπή στην επόμενη συνεδρίασή μας τον Φεβρουάριο. Αντιπροσωπεία στην Ινδία. Παρουσίαση της έκθεσης από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας, τον συνάδελφο Ζαλεύσκη αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σύντομα συμπεράσματα από την επίσκεψή μας στην Ινδία. που έγινε πριν από μερικούς μήνες. Κύριος στόχος μας ήταν να πάρουμε πρώτο χέρι πληροφόρηση από την Ινδική κυβέρνηση το Κοινοβούλιο, εκπροσώπους ε, διαφόρων φορέων και οικονομικών ε, εκπροσώπων και την κοινωνία των πολιτών για ε, τα εμπόδια που υπάρχουν ακόμη για να υπάρξει συμφωνία ελευθερού εμπορίου με την Ινδία δεύτερον για τη θέση της, για τον τελικό γύρο των διπραγματεύσεων για την ένατη συνάντηση, υπουργική συνάντηση του ΠΟΕ στο Μπαλί και την οικονομική και πολιτική πραγματικότητα στη χώρα που επηρεάζει την ε, εμπορική πολιτική της Ινδίας. Καλή ευκαιρία για να τους ενημερώσουμε για τις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια ενδεχόμενη τέτοια συμφωνία εμπορίου με την Ινδία και για την εργασία του ΠΟΕ. Είχαμε ε, πολύ εκτεταμένο πρόγραμμα. Επισκεφτήκαμε όχι μόνο την πολιτική πρωτεύουσα της Ινδίας, το Δελχή, αλλά και την οικονομική και χρηματοπιστωτική πρωτεύουσα της χώρας, την ε, ε Βομβάη, το Μουμπάι και επίσης και το κέντρο της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Πούνα. Ιδίως στην Πούνα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κατάσταση για να καταλάβουμε τις δύσκολες ειδήσεις που αφορούν τους δασμούς για τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά τους, γιατί ήρθαμε σε επαφή με έναν από τους ε, σημαντικότερους παραγωγούς ε, στον κλάδο αυτό Ινδούς αλλά και Ευρωπαίους. Αντιμετωπίσαμε τις δυσχέρειες λοιπόν, ε, καταλάβαμε τις δυσχέρειες ε, που αντιμετωπίζει ο κλάδος γιατί υπάρχει κρίση στον κλάδο αυτό στην Ινδία. Στο Δελχή κάναμε πολύ καρποφόρες, μακρές και έντονες συζητήσεις με τον Λόξ που είναι εκπρόσωπος της, του, της οικονομικής ζωής της Ινδίας, του Κοινοβουλίου. Συγγνώμη. Επίσης συζητήσαμε με την Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας του Κοινοβουλίου και καταλάβαμε καλύτερα τις ανησυχίες ε, που εκφράζονται στην Ινδία σε σχέση με μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Επιπλέον η συμφωνία μας επέτρεψε να αντιμετωπίσουμε κάποιες παρανοήσεις για την Ένωση, τις, πολιτικές της και την Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου. Μας έδωσε επίσης την ευκαιρία η επίσκεψη στο Δελχή, να κάνουμε διάλογο με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών για να διαπιστώσουμε πόσο ζωντανή και ενεργός είναι η κοινωνία των πολιτών στη σημερινή Ινδία. Συζητήσαμε θέματα όπως η καταπολέμηση της εργασίας των νέων, η πρόσβαση στα ε, φάρμακα, η επιστηστική ασφάλεια ανάπτυξη της υπαίθρου και η πνευματική διοκτησία. Επίσης, ε, κάναμε μια συνέντευξη τύπου Οπότε υπήρχε κάποιο αντίκτυπο στον τύπο τη επισκέψή μα. Στο Μουμπάι συζητήσαμε εκπροσώπου των επιχειρήσεων, αλλά όχι μόνο ειδικών, αλλά και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ε, για να ακούσουμε τι θέσει του για μια τέτοια συμφωνία και γενικότερα για τι εμπορικέ σχέσει Ένωσης Ένωση-Ινδία. Οι περισσότεροι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου έχουν επιφυλακτική ε, προσέγγιση έναντι μια τέτοια συμφωνία, αλλά ο το τομέας και ο τομέας ενδυμάτων είναι ιδιαίτερος ε, θετική έναντι μια τέτοια συμφωνίας. Ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα και με το θέμα της πρόβασης στα φάρμακα. Είναι ένα θέμα που το κοινοβούλιο μας ε, παρακολουθεί ε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις διαπραγματεύσεις με την Ινδία. Στις συζητήσεις στην Ινδία διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για το πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις. Ήξεραν λιγότερα από εμά. Γιατί εμείς έχουμε την δική μας ομάδα παρακολούθησης, την δική μας εποπτική ομάδα που παρακολουθεί τις διαπραγματεύσεις με την Ινδία. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους δεν είναι πολύ γνωστή η Ένωση στην Ινδία, ούτε ο ρόλος της και ιδιαίτερα ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι ευρέως κατανοητός από ε, την οικονομική και πολιτική ελίτ της Ινδίας. Η επίσκεψή μας ε, βοήθησε να καταλάβει να καταλάβουν οι συνομιλητές μας στην Ινδία ότι ναι θέλουμε να υπάρξει τέτοια συμφωνία ελευθερού εμπορίου οι διαπραγματεύσει ε, ήδη έχουν διαρκέσει 6 χρόνια, πάνω από έξι χρόνια, αλλά είναι επίσης σαφές ότι δεν είναι πολύ πιθανό να υπάρξει πολιτική συμφωνία πριν από τις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές που θα γίνουν το Μάιο. Η κυβέρνηση είναι συνασπισμός ε, με κύριο εταίρο το κόμμα του Κογκρέσου, αλλά έχει χάσει διάφορες εκλογές σε διάφορες πολιτείες ε, της Ινδίας, σε διάφορα μόσπονδα κράτη και μάλιστα με... Ε, ήταν πολύ βαριές αυτές οι ήττες, ε, βαρύτερες από ό,τι αναμενόταν. Άρα η κυβέρνηση ήδη θεωρείται ότι βαίνει προς το τέλος της. Αλλά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα μπορούσε να επηρεάσει τις ε, διαπραγματεύσεις. Σε τι βαθμό όμως δεν ξέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Μαρία Παντία, που δεν είναι μόνο μέλος αντιπροσωπείας, αλλά είναι και μόνο εισηγήτρια για την Ινδία. Η Μαρία. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με τις ευρύτατες ε, εξής που μας έδωσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπής κ. Ζαλεύσκη. Θα ήθελα να προσθέσω τρία-τέσσερα ε, στοιχεία, δικές μου εντυπώσεις, νομίζω όμως ότι τις συμμερίζονται και οι υπόλοιποι. Αν θυμάστε, για να ξεκινήσω, όταν αξιολογήσαμε τη σκοπιμότητα της επίσκεψης αυτή στην Ινδία, ακριβώς λόγω της κατάστασης ότι θα έχουμε εκλογές και στην Ινδία και στο Ευρωκοινοβούλιο φέτος. Ε, εγώ νομίζω όμως ήταν καλή απόφαση που λάβαμε, επισκεφτήκαμε την Ινδία για να διαπιστώσουμε ποια είναι η διάθεση. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον να, να συνεχίσουν να επεξεργάζονται αυτή τη συμφωνία, ναι ή όχι. Και εγώ νομίζω ότι καλή διάθεση υπάρχει. Όπως υπόθηκε όμως, διαπιστώνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε συμφωνία πριν τις εκλογές. Επίσης, διαπιστώσαμε την ανάγκη να εστιάσουμε ε, στην διαφύλαξη της πρόοδου που έχουμε επιτελέσει μέχρι στιγμής στις διαπραγματεύσεις και στο έτερο συμβαλόμενο μέρος, την Ινδία, θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε δεσμευμένοι απέναντι σε αυτή τη στρατηγική σημασία εμπορική συμφωνία. Βέβαια, ε, λείπουν ακόμη διάφορα ε, θέματα, δεν έχουν ικανοποιηθεί κατέρωθεν απαιτήσει. Επίσης, κάτι που πρέπει να γίνει κατά την άποψή μου είναι να βελτιωθεί η ενημέρωση από την Ινδία για τους εμπλεκόμενους φορείς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, μέσα ενημέρωση, επιχειρηματίες και βουλευτές. Διότι μας δόθηκε εντύπωση ότι δεν είναι σε βάθος γνωστά ε, τα όσα διακυβεύονται οι προκλήσεις ή τι μπορεί να κερδίσει η Ινδία και όχι μόνο αλλά κυρίως η Ινδία αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά, ήταν ενδιαφέρουσα η επίσκεψη. Ξεκαθαρίσαμε τις δικές μας προθέσεις ε, και τις κόκκινες γραμμές που βάζουμε και πρέπει πλέον να περιμένουμε και από την προσεχή κυβέρνηση της Ινδίας αλλά και από την ε, επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδείξουν το ίδιο ενδιαφέρον για να έρθουμε σε ένα αίσιο, να έχουμε αίσια έκβαση. Ναι, να έχουμε happy end. Για να δούμε, μακάρι. Ποιος ξέρει. Ευχαριστώ πολύ για την αναφορά αυτή της ε, αποστολή στην Ινδία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πει κάτι. Σε σχέση με την κατάσταση στην Ινδία, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πώς λέγεστε, για να γραφεί τα πρακτικά. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι εμεί ε, καλωσορίζουμε το ενδιαφέρον που δείχνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη, για τι εμπορικέ σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Ινδία. Ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η επίσκεψη, συνεισέφερε στην ε, προβολή ε, των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Ινδία και του ρόλου που διδραματίζουν τα διάφορα θεσμικά όργανα στην εμπορική πολιτική. Όπω προαναφέρθηκε, οι γενικές δράσεις αναμένονται, μάλλον οι εκλογές αναμένονται τον Απρίλιο-Μάιο στην Ινδία και θα επηρεάσουν σίγουρα τα πράγματα. Εμείς βλέπουμε και από την κυβέρνηση να συνεχίζει τη διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία Ελευθερομπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας. Πρόεδρος, μακάρι. Σημείο 25. της υποπτικών ομάδων. Χιλή. Κυρία Κορέα, η μόνιμη συγκέντρια από το ΕΛΚ. Συγχρονισμός επίσης εμπορικών συμφωνιών με Χιλή και Ινδία. Είναι ένα θέμα που το συζητήσαμε στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της Ολομέλειας. Γι' αυτό το ενδεχόμενο είπα, υποπτική ομάδα, συνεδρίασε στις 7 Ιανουαρίου, ενημερώθηκε από τον Ιγνάθιο Γκαρσία, τον επικεφαλής της διαπραγμάτευσης, για τον τρίτο γύρο των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν ε, στην Ουάσιγκτον το Δεκέμβριο. Είμαι εγώ ο μόνιμος ηγητής, οπότε θα σας πω τι συμφωνήσαμε, ποιο είναι το νέο σχήμα που συμφωνήσαμε με την Κομισιόν. Είπαμε ότι πριν και αμέσως μετά κάθε γύρο θα έχουμε κάποια συνεδρίες. Και αυτό λειτουργεί πολύ καλά ως σχήμα, υπάρχει πολύ καλή ροή ενημέρωσης από την πλευρά της Κομισιόν. ενημερωθήκαμε ότι έχουμε πλέον εντοπίσει τα κοινά σημεία και τις διαφορές. Θα έχουμε ένα πολιτικό απολογισμό μεταξύ Επιτρόπου Ντεχούχτ και Μάικ Φρέμαν σε καμιά δύο-τρεις εβδομάδες. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να σημειώσουμε πραγματική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Για το Μαγρέμπ, Μαγρέμπ η εποπτική ομάδα συνεδρίασης 17 Δεκεμβρίου με εκπροσώπους από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Άγκρη για τη συμφωνία την εμπορική με το Μαρόκο και συζητήθηκε ιδίως το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων. Μαρία Σαρνέζ από την ομάδα Άλντε είναι η μόνιμη σχέτρα, όμως δεν είναι παρούσα. Α, δεν σας είδα. Κρύβεστε γι' αυτό. Come back to Chile. Ας επανέλθουμε στη Χιλή. Δίνω το λόγο στην μόνιμη εισηγήτριά μας. Κρυβόσασταν πριν πίσω από το πίνακα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να σας πω, όπως είπατε και εσείς, ότι την περασμένη εβδομάδα όντως υποβάλαμε μια προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για την εξυγχωρισμού των ε, εμπορικών και συναφών κεφαλαίων στη Συμφωνία Σύνδεσης Ένωσης με Χιλή και με Μεξικό. Για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσα να μετάσχω στη συζήτηση που είχαμε στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα ως μέλος ωστόσο της επιτροπή Παρακολούθησης των σχέσεων με την Χιλή θέλω να σας ενημερώσω για τα σημαντικότερα σε ό,τι αφορά τις προοπτικές εξυγχρονισμού και επικαιροποίησης της Εμπορικής Συμφωνίας Ένωσης Χιλής. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπογραμμίστηκε η επιτυχία της συμφωνίας αυτής από την θέση της σε ισχύ από την 1η Δευτέρα του 2003 ε, καθότι οδήγησε σε αύξηση του διμερούς εμπορίου κατά 128% φτάνοντας τα 18,1 δις ευρώ το 2012. Ομοίως υπογραμμίστηκε ο ιδιαίτερος ε, πολιτικός χαρακτήρας ε, της σχέσης αυτής που συνάφθηκε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματευόταν συμφωνίες με πολύ, πολύ πιο φιλόδοξες με τη ΣΥΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά. Μόνο και μόνο να σας δώσω κάποια ονόματα. Το ίδιο φορά και τη διαδικασία περιφερειακής ενοποίησης που προκύπτει από την Συμμαχία του Ειρηνικού. Η συμφωνία λοιπόν πρέπει να εξυγχρονιστεί, να ενημερωθεί. Να πούμε επίση ότι ο Επίτροπος Εμπορίου δεν ήταν παρόν κατά τη συζήτηση. Ο Σιμ Κάλλας, ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής, ήταν παρόν και έλαβε το λόγο ανταυτού. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του κ. Κάλλας υπογράμμισε τα αποτελεσματικά ε, τα θετικά αποτελέσματα της συμφωνίας και τα θετικά αποτελέσματα και για τη, τη βούληση των δύο πλευρών να εμβαθύνουν περαιτέρω τις εμπορικές σχέσεις. Επίσης, η Επιτροπή δέχθηκε θετικά την πρόταση ανανέωσης ε, που υπέβαλαν οι αρχές της Χιλής στην προηγούμενη συνάντηση της Επιτροπής ε, Σύνδεσης Χιλής ε, Ένωσης τον Οκτώβριο του 2013 που θα εξεταστεί από την Επιτροπή και από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Από πλευράς της Επιτροπή θεώρησε ότι τομεί που μπορούν να τύχουν ενημέρωση και επικαιροποίηση αφορούν τον τομέα των υπηρεσιών, των κανόνων προέλευση, των επενδύσεων, τι δημόσιε συμβάσει, τα τεχνικά εμπόρια στο εμπόριο, υγειονομικά και φυτογειονομικά μέτρα και βιώσιμη ανάπτυξη. Στα συμπεράσματά της η Επιτροπή υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται μια διαδικασία αξιολόγησης για τις πιθανές μεθόδους εξυγχρονισμού της συμφωνίας και έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία διερευνητικών και τεχνικών συζητήσεων το 2014. Κλείνω πιστεύοντας ότι χάνουμε χρόνο μετά την σύνοδο με τη Χίλη πέρυσι. Καλό είναι λοιπόν να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Ελπίζω στην επόμενη συνάντηση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ένωσης Χιλής που θα γίνει εδώ στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα, στις 23 την Πέμπτη δηλαδή, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Μεξικό. Συζητήθηκε Συζητήθηκαν οι προτάσει εξυγχρονισμού τη ε, συμφωνία με το Μεξικό την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο, μαζί με τι αντίστοιχε συζητήσει για τη Χιλή. Ο εισηγητή μα λείπει. Ήμουν εγώ όμω στη συζήτηση. Και αν θέλετε να σα πω κάποιε παρατηρήσει. Πρώτον, δεν ήταν εκεί ο επίτροπο. Ο κύριος Κάλλας τον αντικατέστησε. Μα Μας είπε η Επιτροπή ότι θέλει να αναπτυχθούν οι σχέσεις εμπορίου και επενδύσεων με το Μεξικό, αλλά όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά και υποσυζήτηση με τους ε, Μεξικανούς συνομιλητές μας. Έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις προσφάτως στο Μεξικό που δημιουργούν ενδιαφέρουσες προοπτικές για την Ένωση ιδιαίτερα για τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια, διαβουλεύσεις γίνονται μεταξύ Επιτροπής και της κυβέρνησης του Μεξικού. Η πρώτη συνάντηση έγινε τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες. Συζητήθηκαν πνευματικά δικαιώματα, κανόνες προέλευσης, διευκόλυνση του εμπορίου, ε, φυτικά, ε, υγειονομικά και φυτο-υγειονομικά και άλλα. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στο Μεξικό, θα αφορά δημόσιες ε, προμήθειες, προστασία των επενδύσεων, ενέργεια, αμυντικά μέτρα για το εμπόριο, ανάπτυξη. Θα κάνουμε μία έκθεση μετά από τις συναντήσεις αυτές για το κοινό μας όραμα Η Επιτροπή θα ξεκινήσει μια διαδικασία αποτίμησης των τρεχουσών εμπορικών σχέσεων με το Μεξικό, θα μελετήσει τον κοινωνικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των σχέσεών μας για να ποσοτικοποιήσουμε τα, τους ε, εναπομένοντες φραγμούς στο εμπόριο για να συμπεριληφθεί σε αυτό το τομέα και ε, το πρόβλημα των κοινωνικό περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η απόφαση της Κομισιόν, αν θα ξεκινήσει το πραγματεύσεις, θα εξαρτηθεί από αυτά τα τρία προαναφερθέντα. Έχουν γίνει διερευνητικές επαφές Η Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης για να υπάρξουν νομικά δεσμευτικές κλίσεις. Ε, Πολύ θετική λοιπόν ήταν η προφορική ερώτηση. Μας ε, επέτρεψε να λάβουμε τι τελευταίε πληροφορίε από την Κομισιόν. Η Κομισιόν δεν έχει πάρει ακόμη απόφαση για το πώ θα τα πάει αυτό το θέμα. Και λογική προσέγγιση είναι πρώτα να γίνουν αυτές οι διερευνητικές ε, διαβουλεύσεις και αυτό το κοινό κείμενο και αυτή η μελέτη για το πώς θα μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε τις σχέσεις μας. Το Μεξικό Βεβαίω έχει πολύ ανοιχτή προσέγγιση για τι εμπορικέ σχέσει όπω και η Χιλή, αλλά το Μεξικό ανήκει και στο ναύτα. Τη Συμφωνία ελευθερών Εμπορίου με τη Βόρεια Αμερική έχουμε καταλήξει στι διαπραγματεύσει μα με τον Καναδά, διαπραγματευόμεθα με τι ΗΠΑ και οι συμφωνίε αυτέ ήταν πολύ πιο φιλόδοξε από αυτά που έχουμε με το με αυτά που προβλέπουμε να έχουμε το Μεξικό. Εφόσον λοιπόν καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις με τις άλλες χώρες μέλη της ΝΑΦΤΑ, λογικό να αναβαθμιστούν οι σχέσεις μας και με το Μεξικό. Πολύ θετικέ λοιπόν οι προοπτικές. Θα συναντηθώ με τον πρέσβη του Μεξικού για να κάνουμε μια αποτίμηση της κατάστασης. Συμφωνώ λοιπόν με αυτά που είπε ο κύριος ε, Ζαλεύσκη. Έχουμε λοιπόν ήδη το μηχανισμό που μας επιτρέπει να έχουμε πληροφόρηση, στοχευμένη πληροφόρηση, συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς, την Κομισιόν και τους ε, ξένους συνομιλητές μας. Αυτές οι προφορικές ερωτήσεις αποδεικνύουν Η σημασία τους, τη χρησιμότητά τους, γιατί έτσι η Επιτροπή μας ε, έχει πολύ καλύτερη ενημέρωση από τους συνομιλητές μας στις χώρες αυτές. Αυτό είναι πολύ θετικό. Έχει σχόλια κομισιόν. Όχι, όχι, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ταϊβάν. Άτυπη συνάντηση έγινε στις 16 Δεκεμβρίου. με το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο για την Ταϊβάν. Ο κύριος Προύς είναι ο μόνιμος συζητητής μας. Δεν είναι εδώ. Λίγη συνεδρίασή μας σε διάφορα, όχι, επόμενη συνεδρίαση το Φεβρουάριο και προχωράμε προς το τέλος της ε, θητείας μας. Ευχαριστώ πολύ.